Ξεκινάμε λοιπόν, άρχεται η συνεδρίαση. Κυρίες και κύριοι, πριν περάσουμε ε, στο πρόγραμμα της Ολλανδικής Προεδρίας, ε, πρέπει να σας θέσω ένα θέμα διαδικαστικό. Φαντάζομαι έχετε ενημερωθεί ότι η διάσκεψη των Προέδρων αποφάσισε την Επιτροπή για Εσωτερικές Υποθέσεις και Αστικές Ελευθερίες να την παρακαλέσει